Καλημέρα σας. Ε, Κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Καλωσορίζω όλους τους βουλευτές. Έχω ε, ανακοίνωση να σας κάνω. Στις 16 Ιουλίου του 2009 υπέβαλα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μια ε, ε, αίτηση άρση ασυλίας ενός βουλευτού. Το 2010 ο πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής με ενημέρωσε ότι δυνάμη του ψηφίσματος του Απριλίου 2009 του Κοινοβουλίου σχετικά με τους κανόνες ασυλίας ε, που ισχύουν στην Πολωνία ε, έκρινε η νομική επιτροπή ότι έτσι αυτή ήταν απαράδεκτη. Άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τώρα η κοινή συζήτηση για 36 εκθέσεις παρακαλώ για την απαλλαγή ε, το έτος 2008. Έκθεση του κυρίου Λιμπεράτσκι, Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα 3 Επιτροπή. Έκθεση κυρία Σάντερ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Η έκθεση του κυρίου Μπαρτ Στάς για Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επτά εκθέσεις στη συνέχεια του κυρίου Τσανέτσκι Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Συμβούλιο, ε, Δικαστήριο, Ελεκτικό Συνέδριο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Ευρωπαίο Ελεγκτή Προστασία Δεδομένων. 26 εκθέσεις έχουμε στη συνέχεια τη κυρίας Βερονίκ Ματιό δεν θα σας διαβάσω αλίμονο ε, τις επικεφαλίδες και των 26. Ε, τις στην ημερήσια διάταξη. 26 επαναλαμβάνω εκθέσεις, 26 εκθέσεις έκανε η κυρία Βερονίκ Ματίν απαλλαγή. Άρχεται η συνεδρίαση. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στους συζητητές. Ο κύριος Γκάγερ πρώτος. Ε, Διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι βλέπω, δεν πέσατε εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνεδρίου στο ημικύκλιο. Τι γίνεται, θα πρέπει να εξηγηθεί αυτή η απουσία. Επίση, από ό,τι βλέπω, δεν είναι κανεί ούτε από το Συμβούλιο